θα μιλήσουν οι πολιτικές ομάδες το, από το ΕΛΚ, κυρία Βότονσκολ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Εκατοστή επέτειος μάλιστα είναι. Ε, μέρα γιορτής έχουμε πετύχει πολλά πράγματα αλλά έχουμε και πολύ δρόμο να καλύψουμε και θα το καταφέρουμε αυτό μόνο αν συνεργαστούν οι άντρες και οι γυναίκες. Η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας είναι ένα σύμβολο αλληλεγγύης προς τις γυναίκες ε, στην Ιφίλιο και ε, πρέπει να πω ότι είναι ζωτικό αυτό την εποχή της κρίσης. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ώστε άντρε και γυναίκες να συνεργαστούν για ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά μας. Μόνο μαζί οι άντρε και οι γυναίκες μπορούν να εξασφαλίσουν ισότητα ενώπιον του νόμου, αλλά και κοινωνική και οικονομική ισότητα. 50% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι οι γυναίκες, αλλά κερδίζουν μόνο το 10% του παγκόσμιου, των παγκόσμιων εισοδημάτων και μόνο 5% είναι ηγέτες, γυναίκες ηγέτες. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι φτωχές γυναίκες. Όλα αυτά πρέπει να βελτιωθούν, αλλά δεν είναι το πρόβλημα μόνο η φτώχεια. Πάμε στην Ασία. Θα δούμε εκεί ότι τα γόρια έχουν πολύ περισσότερη αξία, τους αποδίδεται μεγαλύτερη αξία από ότι στα κορίτσια. Είναι παραγωγικά τα γόρια για τις οικογένειες και τα κορίτσια συχνά απορρίπτονται. Τα γίνονται εκτρώσεις όταν ε, γυναίκες περιμένουν κορίτσι. Λαθρεμπόριο γυναικών. Αυτό είναι μια άλλη τραγωδία. Βιασμοί, πόλεμοι. Υπάρχουν ε, πολιτισμικοί λόγοι κάτω από όλα αυτά και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτούς αν πρόκειται να βελτιώσουμε την κατάσταση των γυναικών. Η καταπίεση των γυναικών και στις μουσουλμανικές χώρες για θρησκευτικού λόγους είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Γι' αυτό και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξουμε το ρόλο μας μέσα στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων για να προωθήσουμε την ισότητα μεταξύ γυναικών, ανδρών, κοριτσιών και αγοριών. το, το ζήτημα δεν είναι μόνο η καταπολέμηση της φτώχειας. Πρέπει να απελευθερωθούμε από τις πολιτιστικές προκαταλήψεις. Σημαντικό το έργο της κυρίας Άστον και της Επιτρόπου Τζορτζία Ζαβά σε αυτόν τον τομέα. Αλλά και στην Ευρώπη υπάρχουν ζητήματα. Η πολιτική μας ομάδα με την στήριξη του Τζόζεφ Ντόλ, του Προέδρου μας, ε, θέλει να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια. Ποιο είναι το έργο μας στην Ευρώπη. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την πρόσβαση στην παιδεία για όλους. Δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτό δεδομένο. Πρέπει να αποτελέξει στόχο της στρατηγικής 2020. Ευχαριστώ. Εξ της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών, ο πρόεδρος κύριος Σούλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, μια κοινωνία στην οποία οι άντρες και οι γυναίκες δεν είναι ισότιμοι στην εργασία και στη ζωή δεν μπορεί να είναι μια αξιοπρεπής, μια δημοκρατική κοινωνία. Κύρια προϋπόθεση για δικαιοσύνη στην κοινωνία είναι να χορηγείται άσχετα από το γένος από το φίλο. Για εμά του άνδρες αυτό είναι αυτονόητο. Για τι γυναίκε, όμω ακόμη και στι δικέ μα κοινωνίε, όχι. Και αυτό εκφράζεται ξεκάθαρα σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να εξαλειφθούν το πληγρότερο δυνατόν. Και όπου εμεί ω ε, κοινοβούλιο μπορούμε να συμβάλλουμε σημαντικά. Πού μπορεί η, μια κοινωνία να θεωρεί αυτόν ως ισότιμο εάν για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο άνδρες και γυναίκες πληρώνονται διαφορετικά. Πουθενά δεν φαίνεται η διάκριση κατά των γυναικών στην κοινωνία αυτή κατά τέτοιο τρόπο όπως στον τόπο εργασίας όπου οι γυναίκες κάνουν την ίδια δουλειά όπως οι άντρες και παίρνουν 30-40% λιγότερο μισθό. Αυτή η ντροπή πρέπει να εξαλειφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εάν πρέπει να αποστείλουμε ένα μήνυμα κατά τη διάρκεια διεθνής σήμερα της γυναίκας θα πρέπει να είναι ακριβώς ίσια πληρωμή για άντρες και γυναίκες στον τόπο εργασία. Αυτό είναι ένα κεντρικό αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμείς ε, προσπαθήσαμε να καταβάλει προσπάθειες η Κομισιόν και βλέπω σήμερα τη χάρτα για τα δικαιώματα των γυναικών να προωθείται. Καλό αυτό, το χαιρετίζουμε ευθύ όμω κάπω, και σα παρακαλώ να το μεταβιβάσετε στην κυρία Ρέντινγκ, στον κύριο Μπαρόζο, γιατί θα χαιρόμαστε εάν δεν είχαμε αρκεστεί σε αυτό την προώθηση με μια επίσημη δήλωση, αλλά η αρχική υπόσχεση που είχε δοθεί ότι θα ε, παίξει το ρόλο το κοινοβούλιο, ότι η κοινωνία των πολιτών θα παίξει το ρόλο της να είχαν τηρήσει την υπόσχεση αυτή. Δεν έγινε αυτό, μπορεί όμως ακόμα να γίνει και θα ήμουν ευγνώμονα να μην παραμένουμε σε τέτοιες επίσημες δηλώσεις, αλλά τα θεσμικά όργανα να συνεργαστούν ούτω ώστε αυτό το ένα παράδειγμα που ανέφερα να εξαλειφθεί. Η συνάδελφος Βόρτμαν Κόλ ανέφερε άλλα παραδείγματα, αλλά τη Διεθνή ημέρα της γυναίκας, εμείς οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες θα πρέπει από κοινού να κάνουμε το εξής στην Ήπειρο μας δεν έχουμε ακόμα πετύχει την ισότητα. Αλλά οι δραματικές αδικίες κατά των γυναικών σε άλλες ε, ε είναι φρικτές. Αυτά τα βασικά δικαιώματα των γυναικών και κυρίως των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο που δεν τους δίνονται δεν πρέπει να απασχολούν μόνο στις 8 Μαρτίου. Και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω εκείνους τους πολιτικούς που ασχολούνται με ανθρώπινα δικαιώματα στο σώμα. Κάθε πέμπτη το βράδυ εδώ στο Στρασβούργο συζητιέται το θέμα της παράβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως κατά των γυναικών. Και θα άξιζε το θέμα αυτό πραγματικά τουλάχιστον την παρουσία που έχουμε εδώ σήμερα στο Ινολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νταϊάννα Γόλης τώρα εκ μέρους της ομάδας Άλντε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτή ήταν μια ομιλία που δεν ε, ήξερα ότι θα εκφωνούσα. Μου το είπαν πριν από μερικά λεπτά. Είναι σημαντικό που γιορτάζουμε την επέτειο των γυναικών και ιδιαίτερα είναι σημαντικό που φτάσαμε στην εκατοστή επέτειο από τότε που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία. Θα έπρεπε να είναι γιορτή. Θα έπρεπε να γιορτάζουμε το πόσο έχουν προχωρήσει οι γυναίκες και το πόσο ακόμη ε, πρέπει να ταξιδέψουμε για να φτάσουμε ε, και αναφέρομαι στην ισότητα. Είπατε πρόεδρε ότι θα ήταν ωραίο να έχουμε περισσότερες βουλευτίνες εδώ. Έχουμε βελτιωθεί αλλά δεν επαρκούμε. Και στη Βουλή της χώρας μου υπολογίζουν ότι θα χρειαστούμε 200 χρόνια ε, για να φτάσουμε στην ισότητα στη Βουλή μας με την ταχύτητα με την οποία εξελισσόμαστε. Λοιπόν, τα πράγματα δεν προχωράνε αρκετά γρήγορα για πραγματική ισότητα. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί αυτή τη βδομάδα, το λαθρεμπόριο ανθρώπων και η βία κατά των γυναικών. Την περασμένη εβδομάδα πήγα σε μία έκθεση στην εκλογική μου περιφέρεια, ε, έκθεση ζωγραφικής και φωτογραφιών ε, για γυναίκες που ήταν θύματα λαθρεμπορίου ε, από τη Μολδαβία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες εκτιμήσεις λένε ότι το λαθρομπόριο ανθρώπων ενισχύεται σε αριθμούς. Είναι μεγαλύτερο το εμπόριο αυτό από ότι των σκλάβων της Αφρικής σε 350 χρόνια. Λοιπόν, αν εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό ε, και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τα θύματα αυτού του εμπορίου, πραγματικά θα είναι λυπηρό. Τώρα, υπάρχει και ένα άλλο θέμα ε, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Τα προβλήματα υγείας των γυναικών που, ε, στα οποία δεν αφιερώνουμε το, την ενέργεια που απαιτείται. Πολλά έχουμε να υλοποιήσουμε ακόμη, πολλά μπορούμε να γιορτάσουμε, αλλά μένουν και πολλά να γίνουν. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα εκ μέρους των ε, Πρασίνων, η κυρία Κορνέλισεν. Η 8η Μαρτίου είναι η Παγκόσμια ημέρα γυναικών. Ωραία. Ε, τη γιορτάζω αυτή την ημέρα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Το ίδιο έγινε και με τη μητέρα μου και τη γιαγιά μου. Την 8η Μαρτίου Αισθάνομαι αρκετά απελπισμένη όταν σκέφτομαι όλα όσα πρέπει να γίνουν για να υπάρχουν πραγματικά ίσες ευκαιρίες. Γυναίκες αντιμετωπίζουν βία καθημερινά, φτώχεια επίσης. Πολλές γυναίκες κάνουν τα πάντα για να φροντίσουν τα παιδιά τους και τους γονείς μόνοι τους, μόνες τους. Και τόσο λίγες γυναίκες φτάνουν στα ανώτατα επίπεδα της πολιτικής των πανεπιστημίων, ε, της ε, ε, επιχειρηματικής ζωής. Αλλά όταν σκέφτομαι τη γιαγιά μου που ποτέ δεν μπόρεσε να σπουδάσει και έπρεπε να φροντίσει την οικογένειά της και όταν σκέφτομαι τη μητέρα μου που έπρεπε να αγωνιστεί για να μπορεί να είναι το αφεντικό του εαυτού της αντιλαμβανόμαστε τότε ότι τα πράγματα προχωρούν αλλά προχωρούν μόνο όταν κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Μπορεί βέβαια να συμβάλλει, όχι με λόγια και αοριστολογίες. Ο αγώνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα πάντα συνοδευόταν από όμορφα λόγια. Τώρα λοιπόν έχουμε πληθώρα. Ε, την Παρασκευή η Κομισιόν υπέβαλε ένα χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. Ε, και να ρωτιέμαι γιατί δεν ρωτήσανε την άποψη των ΜΚΟ και του Ευρωκοινοβουλίου πρώτου συντάξουν αυτό το χάρτη, το, τη χάρτα μάλλον. Μου προκαλεί κάποιες ανησυχίες αυτό. Ήταν ένα από τα πρώτα έργα της κυρίας Ρέντινγκ σαν επίτροπος ίσων ευκαιριών και γι' αυτό θα, θα θεωρήσω ότι ήταν καλοπροαίρετο θα ήταν χρήσιμο να έρθει με μια οδηγία κατά της βίας εναντίον των γυναικών, ε, με μια οδηγία για τη γονική άδεια και ε, με άλλα μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν τη συμμετοχή των γυναικών στο χώρο εργασίας ώστε να μπορέσουν να εναρμονίσουν καλύτερα τον οικογενειακό τους χρόνο και τον εργασιακό τους θα ήταν ωραίο να έχουμε ποσοστώσεις όσον αφορά τις ηγετικέ θέσεις στις επιχειρήσεις για γυναίκες. Λοιπόν, αν η Κομισιόν τα ωραία αυτά λόγια τα μετέτρεπε σε έργα, θα ήμουν η πρώτη που θα χειροκροτούσα. Αν θέλουμε αλλαγή, την αλλαγή πρέπει να τη φέρουμε μαζί. Η Κομισιόν, το Συμβούλιο, η δεξιά πλευρά και η αριστερή πλευρά αυτού του Κοινοβουλίου. Η 8η Μαρτίου λοιπόν δεν είναι μόνο η Παγκόσμια ημέρα γυναικών. Είναι και τα γενέθλια του γιού μου. Είναι δύο ετών σήμερα. Δύο ετών έγινε. Ελπίζω γι' αυτόν λοιπόν ότι σε 30 χρόνια η Ευρώπη θα είναι ένας χώρος όπου εκείνος και η γυναίκα του ή ο άντρας του θα μπορέσουν να φροντίζουν από κοινού τα παιδιά τους. Και ελπίζω ότι οι γυναίκες τότε θα μπορούν να έχουν ίσες ευκαιρίες να γίνουν επικεφαλής επιχειρήσεων και να βρουν την ευτυχία. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μαρίνα Γιαννακουδάκη τώρα. Η Παγκόσμια ημέρα των γυναικών μας δίνει μια κοινή ευκαιρία για να επικεντρωθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σήμερα μπορούμε να ασχοληθούμε με τις ε, ανισότητες που αντιμετωπίζουν. Πρέπει να γιορτάσουμε βέβαια και τα επιτεύγματα των γυναικών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο χαιρόμαστε ιδιαίτερα που προχωρήσαμε με τα δικαιώματα των γυναικών. Γυναίκες όπως Emily Parkers, σουφραζέτα, έφερε το δικαίωμα ψήφου άλλη κέρδισε το 1993 το Νόμπελ της Ειρήνης προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. Η Μάργαρετ Θάτσερ, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός, το 1979. Λοιπόν, οι γυναίκες πρέπει να προχωρήσουν ε, εργασιακά και αυτό εξακολουθεί να είναι σημαντικό ζήτημα σήμερα, όπως ήταν και παλιά όταν είχαμε την πρώτη Πρωθυπουργό. Πρέπει να δώσουμε εκπαιδευτικές ευκαιρίες, αλλά δεν φτάνουν. Μπορούμε να νομοθετήσουμε κατά το διακρίσεων στον εργασιακό χώρο, αλλά δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε κατά των πολλαπλών ρόλων της γυναίκας. Σαν, ε, το σαν Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες να έχουν επιλογές. Θέλουν σταδιοδρομία, πρέπει να έχουν την απαραίτητη στήριξη. Θέλουν να μείνουν σπίτι και να ασχοληθούν με την οικογένειά τους. Δεν πρέπει να υποτιμούνται το μόνο νοικοκυρά είναι αυτή, αυτό πρέπει να απαγορευτεί τελείω σαν διατύπωση. Ο καθένας έχει την αξία του ανάλογα με τη συνεισφορά του. Μια ομάδα γυναικών είναι πρώτη σε επιτεύγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιορτάζουμε τη συμβολή τους στις 14 Μαρτίου. Είναι οι μητέρες του κόσμου. Οι μητέρες που εγκαταλείπουν τις φιλοδοξίες τους ανατρέφουν τα παιδιά τους. Με τη σωστή ανατροφή συμβάλλουν στον ίδιο στόχο που έχουμε όλοι. Ισότητα, ανοχή μέσα στην κοινωνία και ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία γίνονται σεβαστά από όλους. Ευχαριστώ. Και τώρα... Η κυρία Μπρίτ Σβένσον έχει το λόγο εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα, πανηγυρίζοντας την ε, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, βλέπουμε ότι εδώ και 50 χρόνια τα Ηνωμένα Έθνη ενέκναν μια κοινή πλατφόρμα. Εκτότε στη Νέα Υόρκη οι υποφαινόμενοι και άλλοι συμμετέχοντες σε αυτή την αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη είδαμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα status κουβό. παρά το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο με την έκθεση ε, ταραμπέλα και άλλα ψηφίσματα, δηλαδή Πεκίνο συν 15, είδαμε ότι τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί. Δυστυχώς οι κυβερνήσεις των ε, ευρωπαϊκών κρατών δεν είχαν υψηλέ φιλοδοξίες για τα δικαιώματα των γυναικών όπως ε, έδειξε το Κοινοβούλιο με τα δικά του ψηφίσματα. Πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι οι κυβερνήσεις των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα του Πεκίνου για να κάνουν κηρύγματα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε κηρύγματα προς τρίτους. Ο πρόεδρος Μπαρόζο πριν διοριστεί υποσχέθηκε την σύνταξη μίας χάρτας για τα δικαιώματα των γυναικών. Σήμερα είδαμε αυτή τη χάρτα και η δική μου ομάδα, η ε, Γκούε, θα πρέπει να εκφράσει την λύπη της για το ε, σχεδόν ε, ανεπαρκές περιεχόμενο αυτού του εγγράφου. Δυστυχώς δεν συμμετείχαν εθνικοί οργανισμοί ή ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές για τη σύνταξη αυτού του εγγράφου και οι ευρωπαίοι πολίτες αποκλείστηκαν από αυτή τη διαδικασία. Κύριε Μπαρόζο, δεν αρκεί μία δήλωση για κοινέ αξίες. Χρειαζόμαστε ένα πολύ ε, εύρωστο έγγραφο όπου να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Θα ήθελα αυτό να είναι το πρώτο προσχέδιο μιας χάρτας υπέρ των δικαιωμάτων γυναικών και μέχρι του χρόνου, μέχρι την επόμενη Παγκόσμια ημέρα γυναικών, να γίνει μια συζήτηση με το Κοινοβούλιο και με τους εθνικούς φορείς καθώς και μη κυβερνητικέ. έτσι ώστε να πανηγυρίσουμε την επόμενη παγκόσμια ημέρα και να δούμε ότι έχει επιτελεστεί πραγματική πρόοδος. Εμείς εργαζόμαστε υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών όλες τις ημέρες, όχι μόνο την 8η Μαρτίου. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Αντρέσεν εξ ονόμης της Ευρώπης της Ελευθερίας και Δημοκρατίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή την ημέρα θα ήθελα όλοι οι πολιτικοί και οι νομοθέτες να σταματήσουν με την έκδοση αυτών των δημαγωγικών νόμων περί ισότητας που κάνουν τη ζωή πιο δύσκολη για τις γυναίκες που επιθυμούν να εργαστούν. Στην ουσία απομακρύνουν τις οργανώσεις από, τους φορείς από να προσλαμβάνουν γυναίκες. Ως εργαζόμενη μητέρα στα 30 χρόνια της επαγγελματικής μου ζωής ποτέ ε, δεν βασίστηκα παρά στα προσόντα και δεν θα ήθελα να τύχω ειδική μεταχείρισης λόγω χρωμοσωμάτων. Όμως έχω συγκεκριμένες απαιτήσει από το Κοινοβούλιο να προωθήσει τις ε, γυναίκες αυτού του κόσμου. Θα ήθελα το πρόβλημα της Ισπανίας να ε, συζητηθεί και να συζητήσουμε και το πρόβλημα πολλών γυναικών και ανδρών που πρέπει να ε, φύγουν από τα σπίτια τους. Θα πρέπει εκεί όπου γίνεται καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να σταματήσει αυτό. Αυτό δεν είναι βία θα ήθελα να προστατεύσετε αυτούς που θέλουν να κοινοποιήσουν τις ανησυχίες τους σε σχέση με τις διαρθρωτικές ανισορροπίες του κοινοτικού προϋπολογισμού, όπως έκανα εγώ 8 χρόνια πριν, για να μην ε, έχουν τη δική μου τύχη. Αυτό δεν είναι βία. Θα ήθελα να είμαστε σαφείς για τον προϋπολογισμό 100% πριν προωθήσουμε αυτή τη χάρτα. Έτσι θα τιμήσετε τις γυναίκες και τους άνδρες της Ευρώπης. Αυτοί που καταβάλλοντας τους φόρους επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει. Η κυρία Μορβάη από τους μη εγγεγραμμένους. Eh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πιστώ την προσοχή των βουλευτών σε κάτι συγκεκριμένο. Είναι μεγάλο σφάλμα να γενικοποιούμε όταν γενικά μιλάμε για τις Ευρωπαίες γυναίκες και τα δικαιώματα των γυναικών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν δεν λαμβάνουμε υπόψη ότι η κατάσταση των, γυναικών, των γυναικών στα μη κράτη-μέλη είναι διαφορετική. Είναι σαν να είναι αυτές οι γυναίκες δεύτερης κατηγορίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προετοιμάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διάφορες εκθέσεις για την κατάσταση των γυναικών στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, γιατί και μέσα στο τουρκό της Ευρώπης υπάρχουν έντονες διακρίσεις εις βάρος των γυναικών. Και <clears throat> ήθελα να τονίσω δύο συγκεκριμένου τομεί που σχετίζονται με την απελευθέρωση, ελεύθερο εμπόριο και ούτω καθεξής. Ο πρώτος τομέας είναι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις αυτές ισχύουν διαφορετικά πρότυπα όσον αφορά την υγεία, τους όρους εργασίας, είτε αναφερόμαστε σε σούπερ μάρκετ, είτε σε υπεραγορές, όσον αφορά παραδείγματο χάρη τα διαλύματα, κατά τη διάρκεια εργασία όσον αφορά τι απολύσεις, ε, όσον αφορά την προσέγγιση κατά τη διάρκεια τη εργασίας. Τα πρώτη λέω, που χρησιμοποιούνται στην Κεντρική Ευρώπη είναι διαφορετικά από εκείνα που χρησιμοποιούνται στη Δυτική Ευρώπη. Και ένας άλλο τομέα είναι η εκτόπιση στο εσωτερικό τη Ευρώπη. Οι γυναίκε αυτέ στην ε, κεντρική Ευρώπη ζουν ε, κάτω από πολύ δύσκολε συνθήκε και έτσι ε, έρχονται στην Δυτική Ευρώπη σαν οικονομικοί πρόσφυγες, εργάζονται σε νοικοκυριά, σαν παραδουλεύτρες, φεύγουν στις πατρίδες τους με τα παιδιά τους και έχουν μια τελείως διαφορετική κατάσταση να αντιμετωπίσουν από ότι οι γυναίκες της Δυτικής Ευρώπης. Η αξιοπρέπειά τους αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Αυτά τα δύο προβλήματα θα πρέπει οπωσδήποτε να τα εξετάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο Τζον Ντάλι και του δίνω και το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, αξιότιμα μέλη. Είναι μεγάλη χαρά για μένα που την πρώτη φορά που είμαι παρόν στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου συζητείται αυτό το σημαντικό θέμα η 8η Μαρτιού που είναι η Παγκόσμια ημέρα των γυναικών. Είναι τιμή για μένα να εκπροσωπώ πίσω την Κομισιό και ειδικότερα την Επίτροπο Ρέντινγκ που θα ηγηθούν της προσπαθίας προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών. Μπορούμε συλλογικά να γιορτάσουμε τα παλιά και τα μελλοντικά και τα σημερινά επιτεύγματα των γυναικών. Πήκε η ισότητα των φίλων στις συνθήκες της Ευρώπης. Ακολούθησαν πάρα πολλά νομικά κείμενα και η νομολογία του δικαστηρίου και υπάρχει πλήρης οπλισμός, αν θέλετε, εξασφάλισης ισότητας στο κοινοτικό επίπεδο. Η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο βασική αρχή, αλλά και προωθητική δύναμη για οικονομική ανάπτυξη. Την περασμένη Παρασκευή ο πρόεδρος της Κομισιόν και η αντιπρόεδρος Ρέτινγκ ανανέωσαν τη δέσμευση της Κομισιόν για την ισότητα των φύλων. Παρουσίασαν τη χάρτα των γυναικών. Η χάρτα των γυναικών είναι η πολιτική δέσμευση της Κομισιόν για να προωθηθεί η ισότητα σε πέντε τομείς. Οικονομική ανάπτυξη, ίση αμοιβή ε, ε, για ίση εργασία, συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων, αξιοπρέπεια, ακαιρεότητα και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Η χάρτα των γυναικών το Σεπτέμβριο του 2010 θα ακολουθηθεί από πλήρη στρατηγική για την εξασφάλιση της ισότητας. Η στρατηγική αυτή θα μετατρέψει τη χάρτα σε πραγματικές δράσεις ε, ώστε να υλοποιηθεί η ισότητα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Είναι φιλόδοξα σχέδια αυτά και βεβαίως η Κομισιόν δεν μπορεί να τα υλοποιήσει μόνη της. Πρέπει να συνεργαστεί με τους βασικούς εταίρους της στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ειδικότερα με εσά το Ευρωκοινοβούλιο και, την... και τις επιτροπές σας η σημερινή ημέρα μας υπενθυμίζει πολύ σωστά τις θεσμεύσεις μας. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και τώρα έχουμε συμπληρώσει τις δηλώσεις, το κατάλογο των δηλώσεων που έγιναν σε σχέση με την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. και σε σχέση βεβαίως με τις συνεχιζόμενες προσπάθειές μας να καταπολέσουμε τη βία και να εξασφαλίσουμε την ισότητα των φύλων. Περνάμε τώρα στο άρθρο 150 παρεμβάσεις διαρκείας ενός λεπτού. Κυρία Μπασέσκο, ένα λεπτό. Προσπαθήσαμε